Αυτό χρειάζεται κάποια εξήγηση που προσπαθώ να σας παρουσιάσω γίνεται πιο απλή. Όταν θα ανοίξει η ψηφοφορία θα δείτε στην οθόνη σας, το έδρανό σας, τα εξής στην οθόνη. Πρώτον, το αντικείμενο της ψηφοφορίας. Τι ψηφίζουμε, εκλογή αντιπροέδρου. Μετά, θα δείτε τον κατάλογο με τα ονόματα των υποψηφίων και τον αριθμό των ελευθέρων ε, θέσεων ακόμα που πρέπει να καλυφθούν αντιπροέδρων. Δηλαδή, θα δείτε εννέα ονόματα υποψηφίων, είναι όμως οχτώ οι θέσεις που πρέπει να καλύψουμε. Αν θέλετε να ψηφίσετε τώρα ένα συνάδελφο ή μία συνάδελφο, μπορείτε να μαρκάρετε το όνομά του ως εξής. Κάτω από την οθόνη σας ε, θα πρέπει να πιέσετε το δεξί κουμπί. Κάτω από την οθόνη έχετε διάφορα κουμπιά. Το δεξί τότε θα δείτε ε, να φωτίζετε το όνομα του υποψηφίου. Αν θέλετε να το ψηφίσετε, θα πρέπει να ψηφίσετε το συν που είναι υπέρ. Είναι το αριστερό κουμπί στη συσκευή ψηφοφορίας. Λοιπόν, για να μαρκάρετε το όνομα, να το δείτε έντονο, θα πατήσετε το δεξί κουμπί κάτω από την οθόνη και για να ψηφίσετε, αν θέλετε να υπερψηφίσετε κάποιον, το συν. Dann leuchtet eine blaue ε, μετά θα ανάψει ένα μπλε φωτάκι, ένα γαλάζιο που είναι για έλεγχο, για να το τσεκάρετε. Και ανάβει γαλάζιο γιατί είναι μυστική ψηφοφορία και δεν βλέπει κανείς πώς ψηφίσατε. Αν ανάψει λοιπόν αυτό το γαλάζιο φωτάκι, βλέπετε ένα αστερίσκο μπροστά από το όνομα που έχετε ψηφίσει. Αυτό σημαίνει ότι αν ψηφίσετε κάποιον θα δείτε στο όνομά του αριστερά έναν αστερίσκο. Και αυτό σημαίνει ότι είναι έγκυρη η εκλογή και τον έχετε ψηφίσει. Για να παραμείνει μυστική ψηφοφορία και να μην δει κανεί ποιον ψηφίσατε, και αν θέλετε να ανεβείτε να κατεβείτε στον κατάλογο ξανά, μπορείτε να το κάνετε με ένα κέρσορα. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας και να ανεβοκατεβαίνει πάντα με το δεξί κουμπί ο κατάλογος για το εκάστοτε όνομα και μπορείτε αυτό να το μετακινείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Και μόλις ψηφίσετε θα, θα εμφανιστεί και πάλι ο δίπλα στο όνομα. Μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίζετε. Μέχρι να πω ότι λύγει Πάνω κάτω τη λίστα τα ονόματα και να ψηφίζετε. Μόνο αυτή τη στιγμή πω ότι κλείνει η ε, ψηφοφορία δεν μπορείτε να πιέσετε το συν ή να ακυρώσετε, να αλλάξετε την ψήφο σας. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική πρώτα ψηφοφορία για να δούμε πώς λειτουργεί. Ακριβώς και να μπορέσουμε να τσεκάρουμε εάν ε, όλοι ε, έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο που ψηφίζουμε. Παρακαλώ και πάλι τους τεχνικούς να μας πούνε αν τα εξήγησα όλα σωστά. Όλα σωστά τα είπα. Ωραία. Πού είναι αυτός ο κέρσορας στο πάνω κάτω. Ωραία. Το βλέπουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα εμφανίζονται ονόματα διαφόρων λαϊκών αειδών. Πλάσιντο Ντομίνγκο, ε, Μονσεράτ Καμπαγιέ, Τζέσι Νόρμα, Λουτσιάνο Παβαρότη, Πλάσιντο Ντομίνγκο, διάφοροι τραγουδιστές της όπερας. Θα κάνουμε μία ε, ψηφοφορία τώρα δοκιμαστική ε, με αυτούς τους λυρικούς αίδους. So, Πρέπει να περιμένουμε ε, λίγο να φτάσουν οι καλλιτέχνες γιατί είναι καθοδόν ακόμα. Ε, κάνουν πρόβες, ζεσταίνουν τη φωνή τους. ο κύριος Παπαρότη δυστυχώς όχι. Bitte noch um einen Moment Geduld, ja. Ένα λεπτό παρακαλώ λίγη υπομονή να κάνουμε. Football players, yeah. Να βάζετε ποδοσφαιριστές καλύτερα λέει κάποιος. Mm -hmm. We could also take former prime ministers. Και πρώην πρωθυπουργούς θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει, γιατί όχι. ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Λάμπερτ. Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν λειτουργεί η δοκιμή. μήπω ε, ε, είναι νέα δική σα συνταγή και δεν μπορούμε εμεί να ξέρουμε για ποιον ψηφίζουμε. Δικό σα τέχνασμα είναι μήπω. Ich warte noch mal Minuten. Περιμένουμε. Πέντε λεπτά. Λυπάμαι λοιπόν, πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί εδώ η τεχνική και τα μηχανήματα. Παρακαλώ λίγη υπομονή κάντε. Euh, λοιπόν, κύριε Λαμπέρ, εξ ονόματος των Πρασίνων, ποιον προτείνετε, τον κύριο Καρέρας. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα και ψηφίζουμε. Να σας εξηγήσω πώς θα... Μάλλον, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Okay. Λοιπόν, ψηφίσατε, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει, εξοικειωθήκατε με το μηχάνημα. Υπάρχει κάποιος που να έχει ερώτηση σε σχέση με το μηχάνημα και την τεχνική λειτουργία. Ξαναρωτώ. Εντάξει, εξοικειωθήκατε όλοι οι συνάδελφοι με το μηχάνημα και τον τρόπο ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας. So, also Λοιπόν, Εψήφισαν 694, 673 έγκυρα, 21 άκυρα, 337 η απόλυτη πλειοψηφία. Δεν εκλέγεται κανένας τραγουδιστής και καμία τραγουδίστρια της όπερας. Λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ακολουθεί τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σας ξαναδιαβάζω τα ονόματα των συναδέλφων που θα ψηφίσουμε. Με αλφαβητική σειρά πρέπει να ψηφίσουμε. Καστάλντο, Κρέτσου, Τσανέσκι, Γκυγιόμ, Λάμστορφ, Λούνατσεκ, Παπαδημούλη, Ρεν και Σασόλη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελπίζω να μπορούμε να ψηφίσουμε. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Bitte sehr, Παρακαλώ κύριε Ερτούκ. Κύριε Πρόεδρε, μία πολύ σύντομη ερώτηση. Κοιτάξτε, σε εμά υπήρξαν κάποιες ε, διαφωνίες. Εάν έχουμε οκτώ Πρέπει να ψηφίσουμε τουλάχιστον πέντε. Όχι, όχι, λέει ο πρόεδρο. Όχι, κοιτάξτε. Μπορείτε να ψηφίσετε ένα μόνο, αλλά κατά το μέγιστο οκτώ. Μπορείτε να ψηφίσετε και κανένα, άμα θέλετε. Ψηφίστε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά ε, κατά το μέγιστο μπορείτε να ψηφίσετε οκτώ. Αλλά έτσι κι αλλιώ οκτώ είναι οι οποίοι θα εκλεγούν. Ναι. Λοιπόν, να σας το διευκρινίσω και πάλι. Έχουμε εννέα υποψηφίους, αλλά οκτώ θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν μπορείτε να ψηφίσετε και τους εννέα, τους οκτώ θα ψηφίσετε. Και ρωτώ πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν συνάδελφοι που ψηφίζουν ακόμα. Από ό,τι φαίνεται ψηφίσατε όλοι. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να ερωτήσω καθαρά επίσημα, ψηφίσατε παρακαλώ όλοι, ολοκληρώσατε την ψηφοφορία. Και επαναλαμβάνω και πάλι, ψηφίσατε όλοι. Κατόπιν τούτου κλείνει η ψηφοφορία. Ψήφισα. 704. 691 έγκυρα ψηφοδέλτια. 13 άκυρα. 346 είναι δική πλειοψηφία. 406 κυρία Κρέτου. Εκλέγεται. Γκυγιόμ. 306. Σασόλη. 394. 384 Ρεν. Λάμπστροφ. Δεν εκλέγεται. Λούνατσεκ 244 δεν εκλέγεται. Τσανέτσκι δεν εκλέγεται. Παπαντιμούλης 210 δεν εκλέγεται. Καστάλντο 115 δεν εκλέγεται. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε και ένα τρίτο γύρο ψηφοφορίας. Και ερωτώ καταρχήν όσους εξελέγησαν Ερωτώ λοιπόν τους εκλεγέντες ε, κατά πόσον συμφωνούν με την εκλογή τους ή υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, ε, συμφωνούν όλοι, εκλέγονται κατόπιν τούτου. Με την ίδια διαδικασία περνάμε στον τρίτο γύρο εκλογής. Θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω ότι στον τρίτο γύρο ισχύει πλέον η απλή πλειοψηφία. Ο κύριος Λούκα. Λούκε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μας εξηγήσετε